Señorías. Κυρίε και κύριοι, εξαντλήσαμε τη μερίσια διάταξή μας. Τα πρακτικά θα σας υποβληθούν στην ε, επόμενη σύνοδο προς έγκριση. Διακόπτουμε. Ε, κύριε Σωτηλίκη, συνεδρίασης.